συζήτηση για το θέμα αυτό της ημερησίας διάταξης και θα ήθελα να σας κάνω δύο ανακοινώσεις από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Μία ανακοίνωση αφορά την αίτηση των Ολλανδικών Αρχών για την άρση της ασυλίας του κ. Κράτσμαν βάσει του άρθρου 2 παράγραφος Αρθού 6 παράγραφος 2 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παραπευθεί αυτή η αίτηση στην νομική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η δεύτερη ανακοίνωση αφορά το γεγονός